Το βράδυ η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο στους διερμηνείς.